Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης που αφορά τη δήλωση της Κομισιόν για την αναπτυξιακή βοήθεια στην Ερυθρέα στο φως των παραδιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν τεκμηριωθεί εκεί. Κύριος Μιμίτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την αναπτυξιακή βοήθεια προ την Ερυθρία βάση τεκμηριωμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει να κάνει με την εξωτερική μα πολιτική και γι' αυτό το συζητάμε συχνά με του εταίρου μα σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένη και τη Ερυθρέα. Το διάλογο αυτό λοιπόν, αλλά και δημόσια, με τι ανησυχίε μα σχετικά με τι παραβιάσει τη Ερυθρέα που δεν τηρεί και δεν προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρειάζονται συγκεκριμένες χειρονομίες. Ελευθέρωση των κρατουμένων που βρίσκονται στο Κομμουνικάντο από το 2001 για παράδειγμα και κυρίως τον κύριο Νταβίτισαν και άλλους ερυθρέους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης τις ανησυχίες αυτές τη θέτει και σε διάφορα φόρα στο Συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για παράδειγμα,